προφορική ερώτηση με ακρό σχετικά με τι αλλαγέ που αφορούν τη θερινή ώρα στην Ευρώπη. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και το λόγο θα λάβει ο κύριο Σβόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, τα ευρήματα της δημόσιας ακρόασης για τις αλλαγές στην ε, θερινή ώρα ε, ήταν σαφή και μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάζει η ώρα γιατί ό,τι, εξοικονομούμε από το φωτισμό το δαπανούμε στην θέρμανση. Το ίδιο βέβαια και για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Ταυτόχρονα 20% των Ευρωπαίων ε, ενοχλούνται, αισθάνονται βαθιά ενόχληση από τις αλλαγές αυτές. 80% δεν αντιλαμβάνονται γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό. Υπάρχουν προβλήματα ε, βιολογικά ε, από τη δυσπεψία, τις αϊπνίες, τις δυσκολίες που φτάνουν όμως μέχρι και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα όπως ε, παχυσαρκία, διαβήτης ή και καρδιακές, προβλήματα. Ιδιαίτερα μπορεί αυτά τα, αυτή η αλλαγή της ώρας να επηρεάζει τα άτομα τα οποία πάσχουν από αυτισμό. 131 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι κοστίζει αυτή η αλλαγή στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαίος πολίτης λοιπόν δαπανά ένα ποσό ισότιμο με αυτό της ε, επιβάρυνσης που έχει για, από την συμβολή του στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να αγοράζει φάρμακα τα οποία χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειε αλλαγή τη θερινή ώρα. Κατά τα άλλα, όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι το θέμα είναι άνευ σημασία και εκείνη ασχολείται μόνο με τα σημαντικά ζητήματα. Είναι, είναι ασήμαντο όντω αυτό το ζήτημα και σε οικονομικού όρου, όπω σα ανέφερα ή σε όρους δημόσιας υγείας που σε τελευταία ανάλυση επιβαρύνουν και, την Ευρωπαϊκή, και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό μπορεί να το χαρακτηρίσει ως όχι σημαντικό ζήτημα, μπορεί τα κράτη-μέλη να μην ε, διαμαρτύρονται. Τα κράτη-μέλη όμως, τα κράτη όμως δεν μπορούν να υποφέρουν από διαβήτη ούτε από κατάθλιψη από κάτι άλλο. Οι πολίτες όμως που υποφέρουν έχουν απευθυνθεί σε εμά και μας έχουν ζητήσει να επιληφθούμε του ζητήματος. Πρέπει να επιληφθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία ζητώ να επαληθεύσει την έρευνα αυτή, έρευνα εννέα πανεπιστημιακών φορέων που μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάζουμε ώρα από το καλοκαίρι στο χειμώνα και αντιθέτως υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μην αλλάζουμε ώρα για να μην βεβαρύνουμε την ε, υγεία των πολιτών. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή των νομικών υποθέσεων και τον πρόεδρο της Πάβελ Σφόμποντα για την ε, τροπολογία αυτή που αναλάβαμε μαζί, Επιτροπή των Μεταφορών και Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, γιατί βέβαια έχει ένα ζήτημα σε σχέση με τα ασφάλεια των μεταφορών, το χώρο των μεταφορών, ε, τις εναέριες μεταφορές, το χρόνο εργασίας, των εργαζομένων μεταφορών και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν κάνει μια κοινή ακρόαση και οι δύο επιτροπές μας ε, στη, για το θέμα αυτό και οι εμπειρογνώμονες μας είπαν ξεκάθαρα ότι αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα αυτής της ε, αλλαγής της ώρας, ενώ είναι αποδεδειγμένες οι δυσμενείς συνέπειες. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα θετικό ε, δεδομένο που να αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή της θερινής ώρας. Συμφωνώ λοιπόν με τα σχόλια του κυρίου Σφόμποντα προς την ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά και κυρίως ε, με την επικρίση για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασχοληθεί σοβαρά με τα ζητήματα αυτά. Το αρχικό επιχείρημα ήταν βέβαια ότι εξοικονομούμε ενέργεια και ως πράσινος αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαι οπωσδήποτε υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ε, αποδεδειγμένο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, αντί να εξοικονομούμε φαίνεται ότι δαπανούμε περισσότερη ενέργεια και αυτό θέλουμε να αλλάξει. Θέλουμε να επαληθευθεί εάν έχει κάποιο νόημα να εμφύσατε το σύστημα όπως έχει τώρα, ιδιαίτερα για το τομέα των μεταφορών όπου σημειώνονται σημαντικά προβλήματα διότι μετά την αλλαγή της ώρας, όταν έχει κοιμηθεί λιγότερο μια ώρα ο πολίτης, αισθάνεται πολύ πιο ε, κουρασμένος, επικίνδυνο λοιπόν για τις μεταφορές. Πρέπει να αλλάξουν ε, τα προγράμματα των τρένων, πρέπει να αλλάξουν τα προγράμματα των αεροπλάνων με βάση την αλλαγή της τελικής ώρας, όσο παλαβό και να σας φαίνεται είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να γίνει βέβαια και η αντίστοιχη προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στο φορέα, της επιμελητίας και ούτε καθεξής στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα γίνεται μια ακριβής καταγραφή των δαπανών. 1,7 δις δολάρια, ε, ευρώ το χρόνο μας κοστίζει αυτό, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι η εξοικονόμηση του, του χρήματος. Θα σας πω εγώ που μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα χρήματα αυτά. Οι πολίτες έχουν προχωρήσει σε πρωτοβουλίε σε διάφορα κράτη-μέλη, μα έχουν αποστείλει επιστολέ σε μένα όπω και στου λοιπού συναδέλφου. Γι' αυτό απευθύνουμε ερώτηση στην Επιτροπή. Γιατί η Επιτροπή απορρίπτει τα επιστημονικά δεδομένα από τι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί δεν τα λαμβάνει υπόψη με σοβαρότητα. Πότε θα γίνει μια νέα διερεύνηση των συνεπειών τη αλλαγή ερηνή ώρα, πού θα υπάρξουν τα δεδομένα για την όποια εξοικονόμηση ενέργεια, πού είναι η αξιολόγηση κόστου και αποτελέσματο, πού είναι η πρόοδη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήση τη ενέργεια που είναι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να καταγράφει η ανακοίνωση της Επιτροπής και ποια είναι η, σχέση, η αναγνώριση μάλλον της σχέσης του πολίτη με τον βουλευτή. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστώ την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και τον κύριο Σβόμποντα και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας κοιτάξτε σοβαρά τα πραγματικά δεδομένα, τα επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπέλτς. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι σε τακτική βάση οι πολίτες ζητούν την κατάργηση της θερινής ώρας, του θερινού ωραρίου. Αμφισβητούν κάποιοι πολίτες ε, τους λόγους για τους οποίους ε, τα κρατημέλη προχώρησαν στη ρύθμιση αυτή. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά τις ανησυχίες των πολιτών, μελετήσαμε προσεκτικά τις διαθέσιμες μελέτες. Οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν ανάμεικτα συμπεράσματα και δεν υπάρχει ένα, ένα κυρίαρχο συμπέρασμα σε σχέση με την <clears throat> εξοικονόμηση ενέργειας, την καλύτερη υγεία κτλ. Ε, τα στοιχεία του οικονομικού ωφέλους ε, ε, από την αλλαγή του ωραρίου ή το θέμα της αύξησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης ηλεκτρικών σκευών, λαμπτήρων κτλ. δεν είναι ισχυρά. Συνεπώς λοιπόν οι ρυθμίσεις του 2001 που βοηθούν στην διασφάλιση της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των χρονοδιαγραμμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση υπάρχει λόγος αναθεώρησης της συγκεκριμένης οδηγίας. Ευχαριστώ. Για τις πολιτικές ομάδες τώρα ο κύριος Ρόιλ, ΕΛΚ. Ο Δύο λεπτά πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Σα εκτιμώ ιδιαίτερος, σα εύχομαι ιδιαίτερος, αλλά είναι ανέδεια, ανέδεια και τίποτα άλλο. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και ανησυχίε, και αν πρέπει να τα λάβετε αυτά υπόψη δεν αρκεί να μα λέτε πάντα καλά ήταν τα πράγματα. Δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση αυτή. Η μελέτη που έχουμε στη διάθεσή μα δείχνει νομίζω ότι που μας παρουσιάσετε εσεί νομίζω ότι είναι απλώ γελία. Απλώς γελία και σε κάθε άλλο θέμα ε, δημόσιας υγείας βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο ε, αντιδρά και αντίστοιχα αντιδράτε και εσείς. Μόνο εδώ πέρα δεν μιλάει κανείς. Και γι' αυτό το κεντρικό ζήτημα κύριε Επίτροπε δεν είναι αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να ανατρέψουμε την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά αν υπάρχει έστω και ένας λόγος να δημιουργούμε τόσα προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων δύο φορές τον χρόνο. Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτή η αλλαγή της ώρας. Εγώ δεν έχω να το αιτιολογήσω αυτό. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έπρεπε να δικαιολογώ κάτι το φυσιολογικό. Γιατί το φυσιολογικό δεν είναι να αλλάζουμε δύο φορέ το χρόνο τα ρολόγια με όλε τι δυσκολίε με όλα τα προβλήματα, με όλη τη δυσφορία. Δώστε μου λοιπόν ένα λόγο, μία απόδειξη γιατί πρέπει δύο φορέ το χρόνο να αλλάζουμε τα ρολόγια και θα είμαι στο πλευρό σα. Ιδάλω. να φύγει αυτή η οδηγία από την κυκλοφορία. Και όπως λέει και η Επιτροπή, λιγότερες διατάξεις. Τι είναι αυτό που λέτε δύο φορές το χρόνο θα αλλάζουμε τα ρολόγια. Έχει κάποιο νόημα να υπάρχει. Αφού δεν υπάρχουν νοήματα, λοιπόν, να καταργηθεί. Προς το παρόν είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε δώσει κανένα λόγο. Προβλήματα μόνο προκύπτουν και ας ξαναγυρίσουμε στην ομαλότητα. Το επιχείρημα για την εσωτερική αγορά είναι το πιο ανόητο από όλα, διότι δεν πρόκειται κανείς, ε, δεν λέμε ότι θα πρέπει στην κάθε χώρα να ισχύουν διαφορετικά ε, συστήματα ή συνθήκες. Αντιθέτως, λέμε βεβαίως, ναι, εσωτερική αγορά και να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά παρακαλώ, και να και το ξεκίνησα, Έχουμε 10.000 υπογραφέ από ανθρώπου που διαμαρτύρονται. Για να μην λέτε ότι άλλοι λένε με ανοησίε. 10.000 να του πάρετε σοβαρά υπόψη. Εκ μέρου Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Ρέκνερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, βλέπετε ότι ξυπνάει πολλά πάθη και ενθουσιασμό αυτή η συζήτηση, έστω και είμαστε λίγοι ε, στην αίθουσα. Βεβαίω είναι ένα ζήτημα πολύ τεχνικό γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την εσωτερική αγορά, έχει να κάνει με την ε, σχέση του χρόνου και του ανθρώπου. Δηλαδή επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου ο βιολογικός του ρυθμός από τον χρόνο και από τις εποχές του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε σε σας έκκληση για την κατάργηση της αλλαγής θερινής χειμερινής ώρας, αυτής της αλλαγής νορολογιών και αυτό το λέω εκ μέρου των ανθρώπων που δεν έχουν ε, δυνατά λόμπι πίσω του, αλλά έχουν ε, τα πιο σοβαρά προβλήματα. Αυτού δηλαδή οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν μεγάλε αποστάσει για να πάνε στη δουλειά του και τα παιδιά του σχολείου. Μα λένε ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξει ο καθημερινό ρυθμό του ανθρώπου και να ξυπνάει πιο νωρί το παιδί για να πάει στο σχολείο. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα μετά τη θέρμανση ή του να φεύγουν από το σχολείο την ώρα που είναι ήδη σκοτάδι. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε του ανθρώπου να δουλεύουν τόσο πολύ, σε τόσο δύσκολε συνθήκε ή τα παιδιά να ξυπνάνε τόσο πολύ νωρί μέσα στο σκοτάδι. Κύλων, ένα, ένα μισή λεπτό κουέ. Ευχαριστώ. Η οδηγία για τη θερινή ώρα Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα πρέπει όμως ε, επιτέλους να παραδεχτούμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή. Αυτό στοιχειοθετείται από τις μελέτες ε, που έχουν γίνει. Ε, το πρόβλημα είναι οξύτερο για τους ηλικιωμένου και για τα παιδιά. Είναι, δυσκολεύονται πάρα πολύ να προσαρμοστούν στην αλλαγή προς τη χειμερινή ώρα. Ε, και μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πνευματικά προβλήματα καθώς και συμπτώματα κατάθλιψης. Δαπανούμε τόσο μεγάλα ποσά και αναρωτιόμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβαρύνει τόσο πολύ τα κράτη-μέλη χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίκρισμα. Επίσης, επηρεάζεται και η οικονομική ζωή με την αλλαγή της ώρας. Θα πρέπει Επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου, στη Ρωσία παραδείγματος χάρη, ξεφορτώθηκαν αυτό το πρόβλημα της αλλαγής ε, της ώρας και τελικά αυτό συνέβαλε στην ευημερία των ανθρώπων και των ζώων. Γιατί εμείς λοιπόν καθυστερούμε, πρέπει να σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι, το άσκοπο παιχνίδι με την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. η χώρα μου μπορεί να είναι στην κεντρική ευρωπαϊκή χώρα. κυρία Χάουταλα. Είναι πραγματικά απίστευτο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει σε μια συνέντευξη τύπου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται μόνο με σοβαρά ζητήματα και ότι αυτό δεν είναι σοβαρό ζήτημα. Είναι απίστευτο που ε, επιδεικνύεται τόση αλαζονία σε σχέση με ανησυχίες των πολιτών στο facebook παραδείγματο χάρη λαμβάνω χιλιάδες σχόλια και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα για τους πολίτες. Το παιδί μου γεννήθηκε το 81 όταν άρχισε αυτή η ιστορία και επηρεάζεται ο φυσιολογικός ρυθμός ύπνου, το βιολογικό ρολόι των ανθρώπων και των ζώων με αυτή την αλλαγή επηρεάζεται όλος ιδιαίτερως η ζωή των παιδιών στην υπηαγωγία, στα σχολεία, επηρεάζεται η κίνηση στους δρόμους, όλα επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή ώρας. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβούμε υπόψη τα όσα έχουν συμβεί από τότε που θεσπίστηκε αυτό το σύστημα, πώς έχει επηρεαστεί η οικονομική ζωή, η ζωή των ανθρώπων και τελικά να καταλάβουμε ποιοι υποστηρίζουν αυτό το σύστημα και όπως είπε και η συνάδελφος γιατί η Ρωσία φροντίζει την ζωή των ανθρώπων και των ζώων και εμείς δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να πω ότι το κόμμα μου έχει θέσει την υπόθεση αυτή εδώ και πέντε χρόνια. Υπάρχουν πλέον βρετανικές έρευνες που λένε ότι ο θερινός χρόνος είναι πολύ καλύτερος για τον άνθρωπο από ότι ο χειμερινός. Ας σταματήσουμε λοιπόν με τον χειμερινό χρόνο. Εμείς επιλέγουμε τον θερινό. Η θερινή ώρα είναι σαφώς προτιμότερη και για εξοικονόμηση ενέργειας Και ξέρετε ότι τίθεται θέμα κατανάλωσης ενέργειας και τα καλοκαίρια πλέον μέσω της χρήσης κλιματιστικών μέσων. Και υπάρχουν και θέματα, στατιστικές μας δείχνουν ότι υπάρχουν θέματα με τους αριθμούς των ατυχημάτων, των οδικών ατυχημάτων. Ευχαριστώ. Μπέκερ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως βλέπετε, εδώ όλες οι πολιτικές ομάδες του σώματος εκφράζουν αποτροπιασμό και αγανάκτηση για την απουσία ε, δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη στάση του Συμβουλίου. Ζητούμε άμεση επαλήθευση της ε, εξαμηνίας αλλαγής της ώρας με επιστημονική, σοβαρή θεμελιωδεμένη επαλήθευση, γιατί αυτά που μας αφηγείστε δεν έχουν καμία αξία και ποιότητα επιστημονικής επαλήθευσης. Εδώ υπολείπεται η Επιτροπή. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με σοβαρά προβλήματα και ως προς το κόστος και ως και κανένα κέρδος σε σχέση με την οικονομία και την ενέργεια. Πολλές πάρα πολλές μελέτες από εννέα δε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια γιατρούς ειδικού που ξεκάθαρα μας λένε ότι προκύπτει τεράστιο κόστος και κίνδυνοι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν δεχόμαστε λοιπόν να μην επαληθεύονται αυτοί οι κίνδυνοι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα σοβαρά στην Ευρώπη. Η μετανάστευση, το ξέρουμε, το ζήτημα των θέσεων εργασία. Αλλά η δημόσια υγεία, η διασπάθηση χρήματο δεν είναι από τα σοβαρά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Βεβαίως και είναι. Και εδώ έχετε μία φωτοτυπία από μια ασφαλιστική εταιρεία της Αυστρίας η οποία καταγράφει με έρθρο της προηγούμενης εβδομάδας 48% περισσότερα τροχαία ατυχήματα με την αλλαγή της ώρας. Δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό. Ο πρόεδρος Γιουνκέρ ε, υποσχέθηκε ότι θα γίνεται επαλήθευση κάθε νομοθετήματος. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει. Παρακαλώ να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να προχωρήσετε σε επαλήθευση και αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε, εδώ και 40 χρόνια οι Ευρωπαίοι δύο φορές το χρόνο αλλάζουν ωράριο. Πρέπει να επανέλθουμε στο ενιαίο ωράριο όπως το έκανε η Ρωσία από το 2011. Οι εμπειρογνώμονε στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2015 δείχνει ότι οι αλλαγές αυτές προκαλούν προβλήματα ε, καρδιακά ε, επεισόδια, προβλήματα ύπνου στους νέους ε, κτλ. Και τα πλέον εκτήματα τα οποία αναμέναμε δεν έχουν επαληθευτεί ούτε μείωση των οδικών ατυχημάτων, ούτε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Θα πρέπει να σταματήσουμε να αλλάζουμε τα ωράρια. Το 76% των Γάλλων θέλουν να διατηρηθεί η θερινή ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει το τι θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Ζαμπόρσκα πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σόμποντα για την επιμονή του και ε, την προσπάθεια που κάνει. Αυτό το διοικητικό μέτρο είναι κάτι που ανήκει στον 20ο αιώνα. Νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε, να σταματούμε επιχειρήματα τα οποία ίσχυαν πριν 100 χρόνια και να δούμε το τι ισχύει σήμερα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αντιμετωπίζει με ηρωνία τις θέσεις του Κοινοβουλίου και αυτό το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, η διοίκηση, δηλαδή ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να έρχεται εδώ να κάνει τον έξυπνο. Δεν είναι αυτή η δουλειά της Επιτροπής και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποβάλει τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε σε εξαντλητική αναλυτική έρευνα. Ο κύριος Φουτζούλικα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα τις σημειώσεις μου στα αγγλικά, αλλά ε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω στα γαλλικά. Αγαπητοί φίλοι, ε, να σας πω ότι τα παιδιά μου πηγαίνουν το κάθε πρωί στο σχολείο και επειδή αλλάζουμε την ώρα, ε, φεύγουν την ώρα που έχει φως. Και εγώ θέλω να πηγαίνουν όταν έχει φως στο σχολείο και να μην ξεκινούν την ημέρα τους μέσα στα σκοτάδια. Βέβαια αυτό ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε με προσεκτικό τρόπο. Υπάρχουν κάποια θετικά. Βλέποντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη με την μετανάστευση, με το ελληνικό χρέος και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, την ανεργία και τα λοιπά και την κοινωνική αναταραχή Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε το θέμα αυτό στην παρούσα φάση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ με ε, την στάση αυτή την περιφρονητική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Μαριάς. Only Greek. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων και το πάθος με το οποίο διεξάγεται η συζήτηση αποδεικνύει ότι πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και νομίζω ο τρόπος με τον οποίο απαντήσατε δεν δείχνει την πρέπουσα σοβαρότητα απέναντι σε αυτό το ζήτημα. καθιερώθηκε η θερινή ώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θεωρήθηκε ότι αυτό είναι κάτι θετικό. όμως βλέπετε ότι οι μελέτες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο διότι έχει γίνει και η δημόσια ακρόαση από πλευράς ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχει αποδειχθεί τεκμηριωμένα πλέον ότι η θερινή ώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία στις μεταφορές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ενώ δεν βοηθάει στη μείωση του κόστους ενέργειας. πρέπει λοιπόν αυτό το σοβαρό ζήτημα να το δείτε να το αντιμετωπίσετε. όταν οι πολίτες ήδη στέλνουν τέτοια μηνύματα ανησυχητικά οφείλει η κομισιόν να κάνει μια σοβαρή μελέτη και να μας δώσει μια σοβαρή απάντηση στο θέμα αυτό. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστώ τους συναδέλφους που κατέθεσαν την προφορική αυτή ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας επισημάνω δεν έναν άλλο τομέα ο οποίος, ε, για τον οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις η αλλαγή της θερινής ώρας. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος πινοκτροφός να εξηγήσει την αγελάδα του ότι άλλαξε το ρολόι. Ξέρετε τι συνέπειες έχει αυτό στη γεωργία. Έχει πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες η αλλαγή της ώρας. Διότι ο βιολογικός ρυθμός δεν αλλάζει. να ακολουθεί η γεωργία, ο αγροτικός τομέας. Και βέβαια ο Γιώργος πρέπει και να πάει το παιδί του στο σχολείο του και να ασχοληθεί με τις αγελάδες του. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία και να τροποποιήσει, να προβήσει την τροποποίηση της ε, ε, οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Στοχოვσκή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν γινόταν σήμερα ψηφοφορία, νομίζω ότι θα σας ζητούσα, Επίτροπε, να μας παραθέσετε τους λόγους ε, για τους οποίους αλλάζουμε την ώρα. Και αν μας δίνατε αντίστοιχες απαντήσεις, ε, πραγματικά θα καταψήφιζα την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ χρειάζομαι και θέλω μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τις ανησυχίες των πολιτών. Εάν τόσα εκατομμύρια λένε ότι θέλουμε να καταργήσουμε αυτό το... Εμ, κατάλοιπο ε, παρελθόντων χρόνων ε, θα ήθελα να λαμβάνετε υπόψη την άποψη αυτών των πολιτών και τις ανησυχίες τους σταματήστε λοιπόν να δείχνετε τόσο ηρωνία και λεζονία για αυτό το ζήτημα. Ας εξετάσουμε σοβαρά το, την επίπτωση αυτών των μέτρων στην υγεία των πολιτών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φων Τι συζήτηση. Βλέπετε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες από τα αριστερά ή μιλάνε, επικροτούν από τα δεξιά, από τα δεξιά μιλάνε, επικροτούν από τα αριστερά δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση. Όλοι θέλουν να καταργηθεί θερινή ώρα, δεν τη θέλουν οι πολίτες και η Επιτροπή. Σηκώνεται και μας λέει δεν έχετε επιχειρήματα. Να, θα λάβετε τώρα το λόγο. Σας παρακαλώ, εσείς τώρα καθίστε και εξηγήστε μας γιατί πρέπει να γίνεται η αλλαγή της ώρας. Εμείς δεν έχουμε να ε, αποδείξουμε τίποτα, ούτε ο πολίτης. Εσείς πρέπει να αποδείξετε γιατί χρειάζεται η αλλαγή της ώρας. Και δώστε μας σοβαρά επιχειρήματα. Γιατί ήταν απλώς ανέδεια αυτά που ακούσαμε πριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου διότι προσδίδουν τη δέουσα σημασία σε αυτό το ζήτημα με διακομματικό τρόπο. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις ανησυχίες. Εσείς εκπροσωπείτε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό ε, σας απευθύνω άμεσα τα ερωτήματά μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους υποβάλλουμε αυτή την προφορική ερώτηση, δηλαδή για, για ποιο λόγο χρειάζεται ε, να αλλάζουμε δύο φορές το χρόνο την ώρα και να επηρεάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ε, δείξουμε ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν ε, με σπουδή να ασχοληθούν με αυτό το τεχνικό ζήτημα και να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών. Να παρακαλούμε να κινητοποιηθείτε και να τροποποιήσετε άμεσα την οδηγία. Ο κύριος Κέλλη, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ από δικές μου παρατηρήσεις ε, τα περασμένα χρόνια είμαι όλο ένα και πιο κατά της αλλαγής της ε, ώρες ε, διότι βλέπω ότι χάνουμε τελικά χρόνο τουλάχιστον ένα μήνα αν υπολογίσουμε την επίπτωση αυτών των μέτρων και μιλώντας για το πώς επηρεάζεται η ζωή των πολιτών και αν το αντισταθμίσουμε με την εξοικονόμηση της ενέργειας βλέπουμε ότι δεν αξίζει 40% περισσότερα ατυχήματα επηρεάζεται η ζωή των παιδιών και τι χρειάζεται να τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδηγία που δεν θα κοστίσει τίποτα και σίγουρα θα είναι οι πολίτες κατευχαριστημένοι και θα δείξετε ότι λαμβάνετε υπόψη τις ανησυχίες του. Και η Ρωσία γιατί το έκανε, γιατί φοβόμαστε να το παραδεχτούμε ότι είχαν δίκιο οι Ρώσοι, διότι είχαν δίκιο και ταχύτατα θα πρέπει ε, να αλλάξουμε αυτή την οδηγία. Θέλουμε όλα να επανέλθουν στο φυσικό βιολογικό του ρυθμό και να μην βγαίνουν στα μαύρα σκοτάδια τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Catch the Eye και τώρα θα ακούσουμε πάλι την Επίτροπο. Κυρία Μπούλτς. Κυρία Μπούλτς, ολοκληρώσαμε την διαδικασία Catch the Eye και σας δίνουμε τον λόγο. Madam President and uh, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Είναι ισχυρότατο το μήνυμα που μου στέλνετε από εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου παρουσίαση, έχουμε επίγνωση ε, των δύο επιχειρηματολογιών υπέρ και κατά του συστήματος. Εγώ προσωπικά συζήτησα με εκπροσώπους πολλών κρατών μελών, τους ζήτησα να μου πούνε την άποψή τους και πρέπει να οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Δεν, είναι, δεν υπάρχει τόση συνέπεια όπως αυτή που ε, διαπιστώνουμε στη σημερινή συζήτηση. Όντως έχουν εκπονηθεί διάφορες μελέτες ε, που ε, μελετούν τον ε, δεχόμενο αντίκτυπο στην υγεία. Όμως δεν προκύπτουν προς το παρόν ε, επιχειρήματα υπέρ ή κατά και θα συμφωνήσω ότι η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από, από αυτό που παραδεχόμαστε και πραγματικά λαμβάνω υπόψη αυτά που λέτε. Όμως ε, πιστέψτε με ότι το κίνητρό μου είναι να διατηρήσουμε την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να έχουμε μια ε, απόφαση η οποία θα λαμβάνεται με ομοφωνία σε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο τροποποίησης αυτής της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, εάν προκύψουν ε, νέα τεκμήρια και παρουσιαστεί μια πιο συστημικού τύπου προσέγγιση, προτιθέμεθα να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ.